Τώρα, στην εμπρισή διάταξη, υπάρχει η έκθεση Ετσεβερία, ολοκληρωμένη αγορά, παράδοσης δεμάτων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για 4 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ενιαία ψηφιακή ευρωπαϊκή αγορά είναι μία από τις προτεραιότητες που θέσαμε στη σημερινή θητεία για να ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η θητεία ήταν αυτή της ψηφιακής αφύπνισης της Ευρώπης. Κατά αυτά τα 4,5 έτη κατορθώσαμε ε, για πρώτη φορά να έχουμε ευκαιρία στον ψηφιακό τομέα για να συμπληρωθεί η ενιαία αγορά, για να βγούμε βγούμε από την κρίση προσαρμόζοντας την οικονομία, το εμποριό μας, τις επιχειρήσεις μας και τους καταναλωτές μας στην ψηφιακή εποχή για να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα που αναμφισβήτητα είναι αυτή που έχει πληγεί ε, τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Μία ευκαιρία για να επενεργοποιήσουμε την αγορά εργασίας και μία ευκαιρία για να εντάξουμε τους νέους μας ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Ε, αναπτύξαμε διάφορες πρωτοβουλίες αυτή τη θητεία που αποτέλεσαν ε, μεγάλο βήμα προς ε, την ενοποίηση και παγίωση μιας νέας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη για την προστασία του καταναλωτή. Το να γίνει ψηφιακή αγορά πραγματικότητα ήταν προτεραιότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή η έγκριση εκθέσεων όπως η συμπλήρωση της, η ολοκλήρωση συγγνώμη, Ευρωπαϊκής στο το 2010 η ολοκλήρωση τη ψηφιακή αγοράς ε, που ψηφίστηκε το 2012 ήταν ένας χάρτης ε, πορείας και αυτός ο χάρτης ε, πορείας ε, υιοθετήθηκε μέσω αυτού του Κοινοβουλίου τον περασμένο Ιούλιο καθόλου αυτό τον καιρό η ειδική ομάδα εργασίας για την ενιαία αγορά είχε μηνιαίες συναντήσεις από τη δημιουργία της τον Ιανουάριο του 2012 και τα συμπεράσματα της Επιτροπής αυτή αυτής ε, συμπεριλήφθηκαν στην εν λόγω έκθεση. Τώρα, κλείνουμε αυτό το κύκλο με την έκθεση που θα υποβάλουμε αύριο σε ψηφοφορία. Η διανομή και η παράδοση των αγαθών που έχουν αγοραστεί επιγραμμικά είναι το απόγειο της ε, του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το να έχουμε υπηρεσίες παράδοσης όχι απλώς είναι θεμελιώδες αλλά είναι ένας από τους πυλώνες όπου έγκυται η εμπιστοσύνη τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα πρέπει να έχουμε υπηρεσίες παράδοσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που να επιτρέπουν σε καταναλωτές και σε επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που εμπορεύονται στο διαδίκτυο τα εμπορεύματα να φτάνουν σίγουρα και σε προσιτές τιμές στον καταναλωτή. Έχουμε μία σειρά θεμελιώδων μέτρων και μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν στον τομέα για να βελτιωθεί η φυστάμενη κατάσταση. Αυτά αναφέρονται στην έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω τους δυο συζητητές για την καλή συνεργασία και τη βούλησή τους για να φτάσουμε σε διάφορες συμβαστικές τροπολογίες στους διάφορους τομείς. Και επομένως είχαμε ομόφωνη υιοθέτηση αυτή τη έκθεση στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Και θέλω να προσθέσω ότι ο δρόμο που διατρέξαμε σε αυτή τη θητεία δεν τελειώνει εδώ. Μένουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να συνεχίσουμε να προχωρούμε και πάρα πολλέ προκλήσει ενωπιών μα. Η επόμενη Κομισιόν και το επόμενο Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποτελέσουν μάρτυρε όλων όσων έγιναν σε αυτή τη θητεία και να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν την ενία ψηφική αγορά. Είναι ένα όνειρο που όλοι θέλουμε να ελοπιθεί και θέλω να κλείσω με έναν τρόπο όπω το έχω κάνει τόσες φορέ σε αυτό το οίκο και δεν κουραζόμαι να επαναλαμβάνω ότι η έξοδο από την κρίση έχει και ψηφιακή μορφή. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα για το ΚΑΤΣΔΙ, συνάδελφος Εσάια. Sisämarkkinoiden kasvupotentiaalia κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε την παρουσία βάσει εκτό για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το είδου υπηρεσίε επιμελητία θα είναι σε επίπεδο που θέλουμε για τι ε, ΜΜΕ, για την διανομή και ότι θα έχουμε την, μια τέτοια πολιτική αποδοτική στην πολιτική απασχόληση. Το συζητήσαμε και συνειδητοποίησαμε ότι πρόκειται για ένα κλάδο που αναπτύσσεται ταχαίως και έχουμε εδώ κάποιες ε, εταιρείε οι οποίες θα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο σύνομο. Οπότε, θα πρέπει να δούμε το ότι οι τιμές τις οποίες διαμορφώνουν ε, γίνονται με τέτοιο τρόπο για να αποκλείουν τους ανταγωνιστές τους από την αγορά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Η Πρόεδρος. Grazie. Livrarea mărfurilor achiziționate online a fost identificată ca fiind una dintre primele cinci priorități pentru stimularea διότι η ψηφιακή αγορά είναι μία από τις πέντε προτεραιότητες. Ίδια συνοριακά εμπόδια υπάρχουν για, τους, για το 50% των εμπορών ελληνικής και έναν στους δύο εμ, καταναλωτές λένε ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στις διασυνοριακές συναλλαγές. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και κατάρτισης και ενημέρωση σε ό,τι αφορά τον τρόπο παράδοσης των αγαθών και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι καταναλωτές αν παραδοθούν καθυστερημένα τα αγαθά ή αν δεν παραδοθούν σε καλή κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει και καθολική υπηρεσία για τις μακρινές περιοχές. Θα πρέπει να βελτιώσουμε και το νομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η έχει το λόγο. Ε, πρόεδρε, αγαπητά μέλη, εκ μέρου ε, του κυρίου Μπαρνιέ, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή και επίσης και την Επιτροπή ΙΜΚΟ για την, για την πολύτιμη συμβολή της ε, ε, στην κοινή δράση για την ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Πριν από λίγο καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στόχος είναι να προσαρμοστεί το ε, περιβάλλον offline σε περιβάλλον online και να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες ε, για τους καταναλωτές και τους ε, παρόχους υπηρεσιών. Σε πάρα πολλούς τομείς καταθέσαμε μία σειρά προτάσεων όπως τον εξυγχρονισμό των ηλεκτρονικών πληρωμών, την ουδετερότητα του δικτύου και το copyright. Μία άλλη σημαντική πρωτοβουλία αφορά την παράδοση των πακέτων αυτές οι δραστηριότητες έχουν επιπτώσεις στην ε, καθημερινή μας ζωή. Η παράδοση είναι καθοριστική σημασία για να διευκολύνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Είναι καθοριστικό στοιχείο για να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στους αγοραστές και τους ε, πολιτές. Ε, καταναλωτές υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάρα πολλοί όμως ανακοινώνουν ότι ανησυχούν σχετικά με την παράδοση ε, των ε, ε, πακέτων αποδοτικότητα του συστήματος είναι ένας καθοριστικός παράγων για το μοντέλο αυτό. Όμως πάνω από το 50% θεωρούν τις ε, διασυνοριακές παραδόσεις ένα εμπόριο. Με λίγα λοιπόν λόγια, για να προωθεί περαιτέρω η ε, περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι offline δομές ε, λειτουργούν αποτελεσματικά. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να καλύπτει τις προσδοκίες των των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, ένα σύστημα που λειτουργεί σωστά για να διευκολύνει την καθημερινότητα, ένα σύστημα το οποίο θα προσφέρει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Υπάρχουν ε, πολλά θέματα ε, που πρέπει να ε, εξεταστούν μέχρι το 2012 και έτσι λοιπόν και με βάση αυτά τα οποία αναφέρονται στην έκθεσή σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα χαρτιπορίας το Δεκέμβρη του 2013 όπου αναφέρονται και άλλες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα παραδόσεων όπως και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και ε, το λιανικό εμπόριο. Στον, στον χάρτη αυτό αναφέρονται επίσης ε, ε, οι ρυθμιστικές αρχές σε σχέση με τους ε, καταναλωτές και υπάρχουν τρεις βασικοί στόχοι. Μεγαλύτερη διαφάνεια, ενημέρωση για όλους τους παράγοντες ε, κυρίως για τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλύτερη διαθεσιμότητα, ποιότητα και διαθεσιμότητα λύσεων παράδοσης, ε, προφανώς ε, διασυνοριακών λύσεων καλύτερη διασφάλιση των καταναλωτών όταν κάτι δεν πάει καλά με την παράδοση να υπάρχουν μηχανισμοί αποζημίωσης. Η πάροχοι, ε, οι παράγοντες και οι οργανώσεις καταναλωτών ήδη έχουν ξεκινήσει επικοδομητικές συζητήσεις. Πολλοί παράγοντες έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν λύσεις που ενδέχεται να ανταποκρίνονται καλύτερα στις προσδοκίες η βιομηχανία είναι εκείνη που καθορίζει τις προσπάθειες. Ε, τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν σύντομα για να καλυφθούν οι προσδοκίες. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν περαιτέρω ενέργειες για να καλυφθούν οι ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών. Έτσι ώστε οι καταναλωτές ε, και το λιανικό εμπόριο να έχουν καλύτερες και διαφανείς λύσεις. Και οι συζητήσεις ε, θα πρέπει να αφορούν και τους κοινωνικούς εταίρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διευκολύνει αυτή τη διαδικασία συνεργασίας και θα συμπεριλάβει όλους τους παράγοντες. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Κοινοβούλιο για να ελέγχουμε ε, τα επιτεύγματα κατά τους επόμενους 18 μήνες και για να μπορούμε να δούμε κατά πόσο χρειάζονται περαιτέρω δράσεις. Σας ευχαριστώ πολύ grazie la discussione è chiusa e la votazione ci sarà domani alle ore. Λοιπόν, αύριο η ψηφοφορία θα είναι στις 11.30. Τώρα, περνάμε στην ε, τελευταία έκθεση, στην ημερήσια διάταξη. Νικολάη, μετανάστες που διαθέτουν επίσημα έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ.